Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ε, έχουν υποβάλει αίτημα για άρση ασυλία του κυρίου και Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού διαβιβάζεται το αίτημα αυτό ε, στην αρμόδια νομική επιτροπή ε, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ελευθερία